Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ο συνάδελφος Αλαφράνκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Your micro, please. Ε, Να υπενθυμίσω στο σώμα, κυρία Πρόεδρε, ότι τον Απρίλιο η πολιτική μου ομάδα ζήτησε να μην συζητηθεί τον Απρίλιο. Υπενθυμίζω λοιπόν στο σώμα τον Απρίλιο η πολιτική μου ομάδα ζήτησε να μην συζητηθεί σε αυτή την Ολομέλεια ούτε η συζήτηση ούτε η ψήφιση για το Γουαντάναμο του ψηφίσματος για το Γουαντάναμο διότι ήταν πολύ κοντά στην ε, τρομοκρατική απόπειρα του, της Βοστόνης. Ο κύριος Βόμποτα πρότεινε να γίνει συζήτηση και η ψηφοφορία να γίνει τώρα. Επειδή έγινε λοιπόν συζήτηση κυρία Πρόεδρε και με βάση το άρθρο 122 του κανονισμού ζητάω να ε, μην γίνει συζήτηση γιατί έγινε τον Απρίλιο. Αύριο λοιπόν το Κοινοβούλιο να κάνει μόνο την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος για το Μαντάνα. Με ευχαριστώ. Κύριε Σαλαφράγκα, ε, θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω με βάση τον κανονισμό ότι θα πρέπει η πολιτική σας ομάδα τώρα να αποστείλει σχετικό γραπτό αίτημα στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ώστε να γίνει η ανακοίνωση στις 3 ε, η ώρα το απόγευμα σήμερα και να μπορέσει να διεξαχθεί αύριο η ψηφοφορία. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα στην ε, ε, ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Γκερέιρα, ναι, παρακαλώ. Α, η κυρία Ντεκάιζερ. Oui. Oui, Madame la simple. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήθελα απλώς για να γλιτώσουμε διοικητικές ε, επιπλοκές να πω ότι η συμφωνία μου συμφωνεί απόλυτα με τον κύριο Σαλαφράγκα. Έχει γίνει η συμφωνία. Απλά να γίνει δηλαδή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνη κυρία Ντεκάιζερ. Λοιπόν, η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ε, ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Νταφ σχετικά με την προσθήκη πρωτοκόλου για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία.